Okay, colleagues. Okay, colleagues, I think we can um, make a start if everybody... Συνάδελφοι, να ξεκινήσουμε. Καθίστε, παρακαλώ. Και καταρχά θα ήθελα να σας ε, καλωσορίσω όλους μετά τι θερινέ διακοπέ. Ελπίζω να ήταν ε, ε, όμορφο και χαλαρωτικό το καλοκαίρι σα. Ελπίζω να μην αισθάνεστε ε, σαν να μην έχετε φύγει ποτέ για διακοπές. Ελπίζω λοιπόν να απολαύσατε το θερινό διάλειμμα και προς τους Γερμηνείς είναι γενικά το λόγο η Πρόεδρος. Είναι η πρώτη συνάντηση της Επιτροπής ε, ΔΕΒΕ, της Επιτροπής Ανάπτυξης, τη νέα σχολική χρονιά αν θέλετε. Και θα είναι μάλλον σύντομη η συνεδρίασή μας. Βασικό σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η ψηφοφορία επί του προϋπολογισμού και επί του ψηφίσματος για το κλίμα. Το πρώτο θέμα λοιπόν στην ημερήσια διάταξη είναι η έγκριση της ατζέντα της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν έχετε αντιρρήσεις, εγκρίνεται. Ευχαριστώ. Κάποιες παρατηρήσεις και ανακοινώσεις μάλλον, πρωτού περάσουμε στις ψηφοφορίες. Ξέρουμε ότι είναι το Ευρωπαϊκό Έτος Ανάπτυξης καταρχάς. Και έχουμε ένα φυλάδιο το οποίο το έχουν καταρτήσει από την ε, Γενική Διευθύνση Επικοινωνίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το Ευρωπαϊκό Αυτό Έτος Το έχετε μπροστά σας. Το έχουμε σε όλες τις επίσημες γλώσσες, σε μεγάλες ποσότητες, στο γραφείο διανομής στον τρίτο όροφο. Από την άλλη πλευρά, δηλαδή μόλις παράσετε τη γέφυρα, του Κωνσταντίνος Καραμαλής, μπορείτε να βρείτε όσα βλάδια θέλετε στη γλώσσα σας. Ε, μόνο στα Λουξεμβουργέζικα δεν το έχουμε. Αν χρειάζεστε φυλάδια για να τα πάρετε για τις εκλογικές σας περιφέρειες. Επίσης, το τελευταίο φυλάδιο για το ευρωπαϊκό, την ευρωπαϊκό θέμα που είναι η ανάπτυξη, της ανάπτυξης μάλλον που είναι η δημοκρατία και η μετανάστευση για το Σεπτέμβριο. Έχετε και στα αγγλικά και σε PDF το κείμενο, όπως συνήθως. Μπορείτε να το βρείτε στο διαθεσμικό, στην διαθεσμική ιστοσελίδα. Η κρίση με τους πρόσφυγες ασφαλώς ε, είναι ένα θέμα το οποίο μα απασχολεί όλου σε όλα τα θέματα. Και η προσωπική μου άποψη είναι ότι θα έπρεπε να έχουμε κάνει πιο πολλά πράγματα και θα πρέπει να κάνουμε πιο πολλά πράγματα. Έχουμε δει και στο παρελθόν ασφαλώ μεταναστευτικέ ροέ, αλλά δεδομένου του γεγονότο ότι πολλοί συνάδελφοι στρέφονται προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ρωτούν τι συμβαίνει με τη σχετική πολιτική. Ζήτησε από τη Γενική Διεύθυνση ΕΚΟ να έρθει και να μας εξηγήσει τι γίνεται με τα θέματα όλα αυτά που άπτονται της αντιμετώπισης της κρίσης των προσφύγων. 21-23 Σεπτεμβρίου στην συνάντησή μας, στη συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Ελπίζω να συμφωνούν οι συνάδελφοι. Επίσης, να πω το εξή. πριν το καλοκαίρι, οι συντονιστέ ζήτησαν να μεταφέρουμε ένα θέμα στην ημερήσια διάταξη τη Ολομέλεια για το Σεπτέμβριο για τα SDGs, για τους ε, βιώσιμους ε, στόχους, ε, αναπτυξιακούς στόχους και τη σχετική διάσκεψη που θα γίνει στη Νέα Υόρκη, με και αποστολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πάρα πολύ σημαντικό ασφαλώς αυτό. Θα γίνει λοιπόν μια δήλωση στην δεύτερη ολομελία του Συμβουλίου. Δεν ξέρουμε πότε ακριβώς. Νομίζουμε όμως ότι θα γίνει την Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου. Και επίση ο Επιτρόπο Δημήτρη δεν θα μπορέσει να παραστεί στι 19 Σεπτεμβρίου στην συναντήση, γιατί θα είναι, στην, θα αλλού. Και προσφέρθηκε να έρθει τη Δευτέρα στην συνεδρίαση μα. Και εκ παραλίλου, προσπαθήσαμε να ενθαρρύνουμε τη συνεργασία με τα Εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προκειμένου να συζητήσουμε πιο εκτεταμένα του ε, βιώσιμου ε, αναπτυξιακούς στόχους και το γερμανικό Bundestag προσφέρθηκε να έρθει να συζητήσει στις Βρυξέλλες ε, τα θέματα αυτά μαζί μας. μας ήρθαν σε επικοινωνία μαζί μας την τελευταία, τις τελευταίες ημέρες πριν τις διακοπές, τον Ιούλιο. Αυτό που προτείνω λοιπόν στην παρούσα φάση είναι να μπουν στην ημερήσια διάταξη, να μπει το θέμα αυτό και να καλέσουμε την ίδια ημέρα που θα συζητηθούν οι βιώσιμοι αναπτυξιακοί στόχοι και το γερμανικό Bundestag για να συμμετάσχει στις συζητήσεις μας. Νομίζω ότι και τα εθνικά κοινοβούλια θα πρέπει να ελέγξουν τους βιώσιμους στόχους της χιλιετίας. 21 Σεπτεμβρίου το απόγευμα λοιπόν προβλέπετε αυτό. Αυτά λοιπόν, αυτά είχα ως ανακοινώσεις να σας ε, αναφέρω. Να περάσουμε στις ε, ανακοινώσεις της Επιτροπής, σημείο 3 της Μερίσιας Διάταξης. Της προηγούμενης συνεδρίασης νομίζω είχαμε αναφέρει ότι ο Βίλιαμ Νίελ θα έρθει να, στην Επιτροπή μας και ότι ο Πίτερ Μανκρέικ που ήταν ο σύνδεσμός μας επί χρόνια με την Επιτροπή αλλάζει δουλειά, αλλάζει θέση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο Βίλιαμ Νίελ ήταν να τον αντικαταστήσει, αλλά μεταφέρθηκε τελικά στο γραφείο του Επιτρόπου Βέλετ. Γι' αυτό έχουμε μία άλλη συνάδελφο εδώ. Δεν ξέρω αν έχει ανακοινώσει να κάνει. Σας ευχαριστώ που εξ ονόματος της ε, Επιτροπής μου επιτρέπετε να σας δώσω κάποιες ε, πληροφορίες ε, για το υπόλοιπόμενο πρόγραμμα του 2015 όπως και για το μελλοντικό πρόγραμμα του 2016. Σε αυτό το στάδιο μπορώ να σας πω ότι οι δύο βασικές πρωτοβουλίες του 2016 θα είναι καταρχάς η εφαρμογή της Ατζέντα 2013 για βιώσιμη ανάπτυξη και πρέπει να εξετάσουμε και τις εξωτερικές και εσωτερικές πτυχές του θεματοφυλακίου αυτού μια αναθεώρηση της πολιτικής ανάπτυξης με τις διαδικασίες της ευρείας δημόσιας διαβούλευσης ε, που θα γίνει στο πρώτο εξάμεινο του 2016. Δεύτερη σημαντική πρωτοβουλία θα είναι ο φάκελος παρακολούθησης της Κοτουνού με το κοινό έγγραφο διαβούλευσης του 2015 για την αξιολόγηση, ανάλυση και τις πτυχές ε, για τη μελλοντική διαδικασία που θα εγκριθεί ως το τέλος του 2016. Προβλέπουμε επίσης μια πρωτοβουλία για την αναθεώρηση του τομέα ασφάλειας με την ανάπτυξη δυνατοτήτων από την άνοιξη του 2015. Συνεχίζεται η δουλειά αυτή ε, για την ε, αναθεώρηση του τομέα ασφαλείας για άλλες πρωτοβουλίες. Ακόμα του 2015 υπό τη μορφή εγγράφου εργασίας, εσωτερικού εγγράφου εργασίας για την ισότητα των φύλων, για την μετάβαση των ε, ε, νεαρών κοριτσιών σε γυναίκες με συγκεκριμένους ε, με πτυχές για την πρόοδο σε αυτόν τον τομέα και ένα, ένα πλαίσιο συνολικά που θα παρακολουθεί τις γυναίκες στη μετάβαση αυτή. Επίσης, έχουμε μια πρωτοβουλία που λέγεται Collect More Spend Better για μια πιο συνεπή ε, προσέγγιση στα πλαίσια των ε, PCD και την ανάπτυξη των προφίλ και της ε, επιφάνειας της εργασίας που γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το έγγραφο εργασία θα παράσχει στην Κομισιόν τη δυνατότητα να προωθήσει νέε πρωτοβουλίε ε, η καταπολέμηση ε, τη ε, μη ένομη χρηματοδότηση και υποστήριξης προ τρίτε χώρες. Τρίτο ή τέταρτο τρίμηνο του 2015 δηλαδή ακόμα φέτο. Επίση προβλέπουμε δημοσίευση για, μέχρι το τέλο του έτου των πληροφοριών ε, των ευρωπαϊκών αποτελεσμάτων, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών αποτελεσμάτων, στα πλαίσια της ετήσιας ε, ανάλυσης αντικτύπου, η δημοσίευση που αναμένεται, όπως έλεγα, για φέτος και τέλος για το 2016, στις αρχές του 2016, η δεύτερη διετής έκθεση για την εφαρμογή του Food and Nutrition τη σχετική ε, πολιτική και πρωτοβουλία, σχετικά με την αποτελεσματικότητα των ευρωπαϊκών παρεμβάσεων και την παρακολούθηση της υλοποίησης των σχετικών έργων και των δεσμεύσεων που έχουμε προς το πρόγραμμα αυτό. Αυτό για το πρώτο τμήμα του 2016 και με την τελευταία αυτή ανακοίνωση ολοκλήρωσα. Σα ευχαριστώ Πρόεδρε ε, χρήσιμες πληροφορίες. Ε, θα μπορούσαμε ίσως να τις αποστείλουμε στους ε, συναδέλφους ε, γραπτός αν τις έχετε κι εσείς. Ο κύριος Γκέρενς έχει το λόγο. Ναι, αυτό ακριβώς ήθελα να ρωτήσω. Με προλάβατε, Πρόεδρε. Να το έχουμε δηλαδή γραπτά. Ωραία. Λέει ο Πρόεδρος. Διάφορες πρωτοβουλίες και εμείς θέλουμε να τις μοιραστούμε με τους συναδέλφους και να έχουμε ενημέρωση στην Επιτροπή νωρί μετά τι διακοπέ. Η ΓΔΕΚΟ έχει επίσης ε, μια ανακοίνωση. Σα ευχαριστώ Πρόεδρε να σα ενημερώσω σύντομα σχετικά με την εχθεσινή επικύρωση μιας ανακοίνωση Towards the World Humanitarian Summit and World Summit for Humanitarian Action. Αυτή είναι ο τίτλος ανακοίνωσης. Η ε, οικοδομή επί τη συνένεση σχετικά με την ανθρωπιστική βοήθεια και τη φιλοδοξία μας ε, για, την, ε, για τον ανασχηματισμό του, του Παγκόσμιου Συστήματος Ανθρωπιστικής Βοήθειας και της ε, σχετικής συνόδου τον ερχόμενο Μάιο στην Κωνσταντινούπολη, όπως και κάποιες συγκεκριμένες συστάσεις που πρόκειται να υιοθετηθούν ή που αναμένεται να υιοθετηθούν, με ευχαρίστως μάλλον να παρουσιάσουμε την ανακοίνωση σε μία από τις ερχόμενες συναντήσεις σας και την παρακολούθησή μας εν ώψη της συνόδου αυτής. Βεβαίω, πολύ σημαντική ανακοίνωση και η Επιτροπή μα θα, θέλαμε, θα ήθελε να έχει μια παρουσίαση. Γνωρίζει ότι ο κύριο Γκέρνιν, ε, μάλλον τώρα καταλαβαίνω δεν ήταν εδώ παρόν σήμερα, αλλά θα είναι σύντομα. Δεν ξέρω αν έχουμε κάποια ερώτηση ή παρατήρηση για τι ανακοινώσει αυτέ. Ευχαριστούμε λοιπόν και θα συνεχίσουμε και εμεί την παρουσίαση των θεμάτων αυτών. Πάμε τώρα στο σημείο 4 που είναι η ψηφοφορία επί της νέας ε, Διεθνούς Κλιματικής Συμφωνίας στο Παρίσι, της ΚΟΠ, που θα είναι πολύ σημαντική αυτή η διεθνής ε, συνεδρίαση, συνάντηση, θα πρέπει να έχει το δικό μας input. Πρωτού ψηφίσουμε, δεν ξέρω κανένα πώς αν η κυρία Ζαμπόσκα θα ήθελε κάτι να πει σχετικά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ήθελα, θα ήθελα απλώς να ευχαριστήσω τους ε, συνεισηγητές ε, και την γραμματεία για την βοήθειά τους και την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε. Ευχαριστώ. Ξέρω πόσο δύσκολο είναι να τα έχουμε αυτά τόσο σύντομα μετά τις διακοπές, γιατί λείπουν αρκετοί. Σας ευχαριστώ για τη δουλειά σας. Πρωτού πάμε στην ψηφοφορία, λέει η Πρόεδρος. Η Γραμματεία θέλει να κάνει μια δοκιμή. Αν θέλετε λοιπόν, πιέστε οποιοδήποτε κουμπί στο μηχάνημα για να δούμε αν δουλεύει καλά το σύστημα ηλεκτρονικής ιοφορίας. Να την κλείσουμε εδώ. Ε, έχουμε ψηφίσει οτιδήποτε, δεν έχει σημασία. Φοβούμαι ότι έχω έρθει χωρίς την κάρτα μου, πρόεδρε. Φοβούμαι ότι την εξέχασα. Θα, θα, θα σηκώνω το χέρι μου αν συμφωνείτε. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε μια υπερβολική ψήφο από τους σοσιαλιστές, βλέπω, λέει η Πρόεδρος. Uh, Αν είναι μόνο ένα μέλος χωρίς κάρτα, θα το προσθέτουμε στον έλεγχο. Αν ήταν περισσότεροι δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό. Για ένα άτομο και μόνο μπορούμε, ελπίζω να μην έχουμε τόσες πολλές οριακές ψήφους, εν So um, we move first then to the, the series of compromises. I'm grateful to να ευχαριστήσω λοιπόν τους ε, συναδέλφους που έκαναν συμβαστικές ε, προτάσεις. Συμβαστική πρόταση 1, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Και περνάμε τώρα στη συμβαστική παριθμών 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά για την συμβαστική 5. Την τροπολογία 9 διορθώνει η Πρόεδρος. Εντάξει, τε λήξη της Εγκρίνεται. Η 12 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 13. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 16. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 21. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. 22 υπέρ. Α, συγγνώμη, 22. Υπέρ, κατά, άποχες, εγκρίνεται. 26 υπέρ, κατά, άποχες, εγκρίνεται. 27 υπέρ, κατά, άποχες, χρειάζεται ηλεκτρονικός έλεγχος για την 27, έναρξη ψηφοφορίας. Πέρασε. Εντάξει, κυρία Πρόεδρε, βρήκα. Ω διαμαγεία βγήκε η κάρτα μου. Μάλιστα, απορρίπτεται γιατί έχουμε ισοψηφία. Απορρίπτεται. 28. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. 29. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Η 30. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 32. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 33. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 36. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Με τις ίδιες πλειοψηφίες. 37 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 39 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 40 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 41 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 42 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 45 στην επόμενη σελίδα. Υπέρ, κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 48. Υπέρ, Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 49. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και περνάμε στη 53. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 56. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 59. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ψηφίσουμε το σύνολο του κειμένου ηλεκτρονικά. Έναρξη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, παρακαλώ. Πέρας. Δεν ψήφοι υπέρ, καμία κατά, δύο αποχές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Ζαμπόφσκα και όλους τους συναδέλφους για την καλή συνεργασία από πλευρά της... Ε, θα το προωθήσουμε αυτό στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Επόμενο θέμα λοιπόν τώρα είναι το 5 της ημερήσιας διατάξης. Ε, θα ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό για να αποστείλουμε την γραμματότησή μας στην Επιτροπή Προϋπολογισμού ασφαλώ. Ο εισηγητής δεν είναι εδώ σήμερα. Δεν έχετε την να πείτε όμως. Να πάμε στη ψηφοφορία λοιπόν κατευθείαν. Δεν έχουμε τροπολογίες εδώ πέρα. Α, έχουμε. Έχουμε πιο, πολύ, πιο μεγάλους αριθμούς όμως. Τα τελευταία δύο ψηφία. 44. Υπέρ κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 45. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 46 <clears throat> υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 57.00 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 5731 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 01 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 02 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 03 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται 04 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 05 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 06 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 07 in favor against 07 εγκρίνεται 36 υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. 26. Όχι, όχι, καταπίπτει 26. Άρα πάμε στην 37, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 09, 09 με συγχωρείτε. Όχι. Μάλλον όχι. Η 10, υπέρ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 Προφορική 1 του εισηγητή. Κυρία Χόιμπρουκ, για την προφορική. Ναι, θα μιλήσω γερμανικά. Μια ερώτηση έχω να κάνω. Είχαμε συμφωνήσει να ψηφίσουμε μόνο τα πληθυκά προγράμματα, τα οποία είχαν συμπεριληφθεί με θετικό πρόσημο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά τώρα συμπεριλαμβάνονται και προγράμματα που είχαν αξιολογηθεί αρνητικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν ε, καταλαβαίνω γιατί πρέπει να τα ψηφίσουμε και αυτά. Ο κύριος Νόιζερ για να απαντήσει. I don't know. I mean, it's on the voting list now. Είναι στο κατάλογο ψηφοφορίας. Μιας και είναι λοιπόν, ας το ψηφίσουμε και όποιον του αρέσει ας το καταψηφίσει. Δεν ε, ήταν θέμα διαδικασίας. Να ψηφίσουμε δηλαδή θα έλεγα. Να ψηφίσουμε, να ψηφίσουμε. Uh, να ενημερώσω απλώς Αυτά είναι τρέχοντα και αυτός είναι ο μόνος λόγος που συμπεριλαμβάνεται. Είναι προφανώς από την προηγούμενη περίοδο της Επιτροπής, λέει η Πρόεδρος. Εν πάση περιπτώσει, ας ψηφίσουμε για την προφορική ένα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Προφορική 2. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 24 υπέρ κατά αποχές Ας ελέγξουμε. Ας ελέγξουμε. Ενέξη προφορίας. Κύριος Νόιζερ, δεν ξέρω γιατί καταψηφίζουμε το συνάδελφο. Δεν είναι στον κατάλογο, βέβαια, αλλά... The vote, is closed. Πέρασε πληροφορία, λέει ο Πρόεδρος. Και εγκρίνεται. Και οι σοσιαλιστές μπορούν να αναρωτιούνται γιατί καταψηφίζουν το συνάδελφο. Λοιπόν, 25 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Προφορική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 51 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 17 <clears throat> υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 19 υπέρ όχι 19, 30 και 40 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται λοιπόν τελική ψήφο δεν έχουμε να ευχαριστήσω λοιπόν τον Άρνε Λίτς ε, και τους συνεισηγητές και μπορούμε να αφήσουμε τώρα το 5 και είναι τέλος της ψηφοφορίας για σήμερα και στο 6 πάμε που είναι η συζήτηση για τον προπολογισμό. Ο Ανελίτς δεν μπορούσε να είναι μαζί μας σήμερα, σήμερα. Ο Νόιζερ αντικαθιστά τον κύριο Λίτσα. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη εξ ονόματος του συναδέλφου Ανελίτς, ο οποίος βρίσκεται στην ε, πόλη του σήμερα, γιατί ε, επισκέπτεται ο Υπουργός ε, κ. Μούλερ την πόλη του. Και είναι, όπως είπαμε, σημαντική αυτή η σύνδεση και με τα εθνικά κοινοβούλια και με τις εθνικές κυβερνήσεις. Με παρακάλεσε λοιπόν να πω δύο λόγια για την τοποθέτησή του, για την γνωμοδότησή του και κάποια σημεία θα ήθελα να τα υπογραμμίσω ιδιαίτερως. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να αποτεχτούμε τις περικοπές του Συμβουλίου. Γι' αυτό λοιπόν οι πιο πολλές τροπολογίες ε, επί του προπολογισμού έχουν να κάνουν με την επαναφορά στα επίπεδα που είχε προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον προπολογισμό. Νομίζω ότι όλοι όσοι παρακολουθούμε τις ειδήσει τις τελευταίες εβδομάδες αλλά και ακόμα τώρα είναι, ξέρουμε ξεκάθαρα πόσο μεγάλη έκτηση έχει η κρίση των προσφύγων. Γι' αυτό λοιπόν θέλουμε κυρίως και στις ε, σχετικές επικεφαλίδες να έχουμε πιο πολλά μέσα για το άσυλο και τους πρόσφυγες για να χρησιμοποιηθούν για μέτρα για να καταπολεμήσουμε τις αιτίε των, των προσφυγικών ροών και για να διοργανωθεί η υποδοχή των ε, προσφύγων στις χώρες. Επίσης, θέλουμε 56 εκατομμύρια ευρώ να δαπανηθούν επιπλέον στον προεπλογισμό για μέτρα εκπαίδευση στα προσφυγικά καταλήματα, για να αποφύγουμε χαμένες γενιές, όπως ονομάζονται, και να υποστηρίξουμε ιδιαίτερα τα παιδιά, τους νέους, που βρίσκονται υποδίωξη και που επί χρόνια δεν έχουν πρόσβαση σε εκπαίδευση. Αυτή ήταν εν συντομία η τοποθέτηση του Ανελίτς και εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί του και θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω και για την καλή συνεργασία με τους άλλους κοιόδησίτες. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Ο λόγο τώρα για τους συναδέλφους από τις ομάδες. Ο κύριος Στήρ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο σκιώτης ηγητής μας, ο Γιώργο Κιμψέρα, δυστυχώς και αυτός δεν μπόρεσε να παρευρεθεί σήμερα. Είναι στη συνάντηση του ΕΛΚ στην Κάτοβιτσε. Εξ του, λοιπόν, θα ήθελα να, συγχωρώ, να συγχαρώ και εγώ τον Ανελής για την γνωμοδότηση αυτή που προετοίμασε. Νομίζω ότι αποστέλει τα μηνύματα που χρειάζεται ακριβώς ιδιαίτερα με το σύνδεσμο που γίνεται, τη σύνδεση που γίνεται μεταξύ της κρίσης των μεταναστών και την ανάγκη αύξησης των πόρων για την αναπτυξιακή συνεργασία στην Ολομέλεια όταν συζητήσαμε το θέμα της κρίσης των μεταναστών. Σε διάφορες περιστάσεις ακούσαμε ότι η αναπτυξιακή πολιτική αποτελεί τμήμα της λύσης. Όταν όμως τα πράγματα φτάνουν στον προϋπολογισμό, τι βλέπουμε, περικοπές. Αυτό δείχνει τεράστια συνέπεια. Σωστό μήνυμα λοιπόν είναι αυτό από πλευράς της Επιτροπής Ανάπτυξης ότι είναι απαράδεκτη αυτή η κατάσταση. Αυτή είναι η βασική γραμμή που διακατέχει τη γνωματότηση και υποστηρίζεται απόλυτα από το ΕΛΚΑ. Και νομίζω ότι επιπλέον το αίτημα να προσταθούν 26 εκατομμύρια για την εκπαίδευση στα προσφυγικά καταλήμματα συνάδει απόλυτα με τις προτεραιότητες που συζητήσαμε πριν το καλοκαίρι. Πάρα πολύ σημαντικό και καλωσορίζω για να μας συμπεριληφθεί αυτή η γραμμή στην γνωμοδότηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Γκέρεντς. Euh, Ευχαριστώ πρόεδρε. Η Κομισιόν από ό,τι φαίνεται έχει διαθέσει ένα δισεκατομμύριο για τη βοήθεια της Αφρικής ε, στο πλαίσιο της ε, παρούσας κρίσης ε, ε, με τους μετανάστες. Η ερώτηση με καταρχάς είναι ακριβή, η ακριβή συμπληροφορία αυτή. Και από πού θα προέλθουν αυτά, από το Ταμείο Ανάπτυξης ή σκοπεύει η σκοπευει η κομισιο να ανοίξει νέο, νέα γραμμή, νέο κονδύλι. Και αυτό θα ξεκινήσει από το 2016 ή μήπως υπολογίζει η μήπω υπολογιζει η κομισιον σε μια συνεισφορά των κρατών μελών που έχουν ιδιαίτερες αμφιβολίες για τις ήδη ανηλυμένες δεσμεύσεις. Θα ζητήσω, λέει η Πρόεδρος από την Κομισιόν, να σχολιάσει στο, τέλος, η κυρία Χόιμπρο και μετά η Κομισιόν. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Άρνελιτς ε, για την έκθεση αυτή. Εμείς από πλευρά των Πρασίνων υποστηρίζουμε απόλυτα το κείμενο και πιστεύουμε και εμείς ότι θέτει τις σωστές αρχές στο κείμενο αυτό. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, προβλέπει πολύ μικρή αύξηση των μέσων, 2% περίπου και δεδομένη της κρίσης πληρωμών που ζήσαμε τα τελευταία χρόνια και η οποία ακόμα δεν έχει προβληθεί αναρωτιόμαστε αν αυτό υπαρκεί και κατά πόσον οι εκκρεμείς λογαριασμοί μπορούν να καλυφθούν με αυτή την αύξηση. Παρ' όλα αυτά λοιπόν το Συμβουλίο θέλει να μειώσει, να περικόψει. Σημαντικά μάλιστα τα μέσα αυτά. Είναι προβληματικό λοιπόν αυτό το οποίο και σωστά πείθεται ως τέτοιο. Και θα ήθελα επίση να υπογραμμίσω αυτά που είπε και ο Ρόμπερτ Νόιζερ αλλά και ο κύριος Στυρ ότι οι περικοπές στον τομέα της μετανάστευσης δεν είναι κάτι αποδεκτό. Σε καιρούς όπου στην Ευρώπη έχουμε πρόσφυγες πιο πολλούς ε, από παρά ποτέ μετά το δεύτερο παγκάσμιο πόλεμο, δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε έτσι. Ούτε θεωρώ ότι είναι αποδεκτό να υπάρχουν οπουδήποτε κοπέ. Βρισκόμαστε σε ένα έτος ανάπτυξης, Παντού ζητάμε αυτό το στόχο το 0,7% τον οποίο και εμείς ήδη δεν καταφέρνουμε να το εκπληρώσουμε. Θα πρέπει να τακτοποιήσουμε το του οίκου μας και να πετύχουμε επιτέλους αυτό το στόχο. Το Συμβούλιο θέλει τουλάχιστον να αυξήσει την ανθρωπιστική βοήθεια. Να την ε, τονίσουμε αυτή την πρόταση. Η προστασία του κλίματος και αυτό βασικό θέμα που μας απασχολεί πολύ ως πράσινος. Και φυσικά καλωσορίζουμε ιδιαίτερα στο γεγονό ότι οι περικοπέ τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, σε ό,τι αφορά το κλίμα ε, ουσιαστικά ακυρώνονται. Αυτό συνάδει με του στόχου μα. Ευχαριστούμε λοιπόν και πάλι την Άρνε Λίτση για την καλή αυτή έκθεση και σα ευχαριστώ όλου που συμφωνούμε για το θέμα τη μετανάσταση και μπορούμε έτσι να συνεχίσουμε τι εργασίε μα. Πουντσολίκα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη αντιμετωπίζουν μια πολύ πολύ δύσκολη κατάσταση αντιμετωπίζοντας αυτά τα ρεύματα μεταναστών που προσέρχονται στην Ευρώπη και το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία για το μέλλον της Ένωσης. Απέναντι λοιπόν σε αυτήν την πολύ σοβαρή πρόκληση η Κομισιόν, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να υιοθετήσουν, σε, να υιοθετήσουν σημαντικότατες αποφάσεις και ίσως έχει έρθει η ώρα να σημάνουμε συναγερμό σχετικά με την απουσία στρατηγικής και την απουσία οράματος από πολλούς από τους ηγέτες μας σχετικά με το μέλλον μας. Γνωρίζετε ότι είμαι ένα από τα μέλη που είναι απολύτως υπέρ της ενίσχυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των θεσμών της γιατί δεν υπάρχει καμία άλλη λύση για την Ευρώπη παρά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γι' αυτό ειλικρινώς δεν κατανοώ με ποιον τρόπο ε, σκοπεύει το Συμβούλιο να περικόψει τους πόρους της ανθρωπιστικής βοήθειας σε αυτές τις στιγμές κρίσης χωρίς προηγούμενο που αντιμετωπίζουμε. Αυτή η τάση θα πρέπει να καταπολεμηθεί πάση θυσία. Και την ίδια στιγμή αρκετοί από τους ηγέτες μας δεν κατανοούν ότι θα πρέπει με κάθε τρόπο να αποκαταστήσουμε να εξισορροπήσουμε την κατάσταση τις περιοχές από τις οποίες έρχονται οι άνθρωποι αυτοί. Βεβαίω και πρέπει να παράσχουμε τρόφιμα και βοήθεια, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αποφασίσει σημαντικά πράγματα σχετικά με την ε, ειρήνευση ή εν πάση περιπτώσει ε, σταθεροποίηση κάποιων περιοχών ή στην ε, εγγύς Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική διότι αν συνεχίσουν έτσι τα πράγματα θα είναι αφόρητα για τους πολίτες, για τις κυβερνήσεις, για τους θεσμούς μας. Κάλλιο αργά παρά ποτέ λέει το γνωμικό. Και ελπίζω το αργά να μην σημαίνει ποτέ. Θα πρέπει νομίζω λοιπόν από κοινού να δώσουμε, να μεταδώσουμε ένα σημαντικό μήνυμα συναγερμού για την ανθρωπιστική βοήθεια και για ασφαλείς περιοχές για όλους αυτούς τους ανθρώπους. Σας ευχαριστώ βεβαίως και θα γίνει σοβαρότητα συζήτηση στο Στρασβούργο την ερχόμενη εβδομάδα για την κρίση αυτή των προσφύγων και θα υπάρξει ψήφισμα όλων των πολιτικών ομάδων ε, σχετικά με την κατεπίγουσα αυτή κατάσταση που πρέπει, έχετε δίκιο να την αντιμετωπίσουμε αυτή τη στιγμή, διότι οι άνθρωποι υποφέρουν τη στιγμή που μιλούμε εδώ. Λοιπόν, δεν βλέπω κάποιο μέλος να ζητάει το λόγο, αλλά έγινε μια συγκεκριμένη ερώτηση από τον κύριο Κιόριν στην Επιτροπή, στην Κομισιόν. Έχουμε γάμα δέλτα ντεύκο και έκο εδώ. Δεν ξέρω ποιος από εσάς θέλει να έχει το λόγο. Καλημέρα σας εκ μέρους της ΔΕΒΚΟ, μονάδα προϋπολογισμού. Δεν μπορώ να... Δεν μπορώ... Μάλλον, υπάρχει πράγματι υπέρ του Σαχέλ ένα ταμείο, η πρόθεση της δημιουργίας ενός ταμείου ενός δις, άνω του ενός δις, και θα είναι ανοιχτό σε δωρητές, δωρητές μεταξύ των οποίων τα κράτη-μέλη. Αν έχετε άλλες ερωτήσεις, μπορώ να σας απαντήσω γραπτός. Η ερώτηση ήταν κατά πόσον προέρχονται αυτά τα χρήματα από τον προϋπολογισμό DEVCO ή από το EDF Κομισιόν. Και τα δύο. Μεγάλο τμήμα από το Ταμείο Ανάπτυξης, αλλά και κονδύλια θεματικά από την ΤΕΠΚΟ. Αλλά θα είναι ένα καταπίστευμα όχι κονδύλι του προϋπολογισμού. Έχουμε και το καταπίστευμα ΜΠΕΚΟΥ, αν ακούσαμε καλά την ομιλήτρια, που είναι και αυτό με συμμετοχή διαφορετικών ε, ταμείων και άλλων ε, εισφορέων και δωρητών. Ο ε, κύριος Γκέρινς. ακούστε, έχουμε μάλλον ένα σοβαρό πρόβλημα επικοινωνίας εδώ. Οι εισφορές έχουν κατέλθει των κρατών μελών, ανακοινώνουμε νέα ταμεία κλείνουμε μία τρύπα για να ανοίξουμε μία άλλη και όλα αυτά σε μία γενικότερη τάση καθόδου και περικοπής των εισφορών και των δαπανών. Δηλαδή θα ήθελα να έχω ένα κατάλογο των υποσχέσεων των κρατών μελών και της πραγματικότητος για να ξεσκεπάσουμε εν πάση αυτή την υποκρισία. Δεν αναφέρομαι μόνο στην ε, Κομισιόν εδώ, αλλά όλο αυτό μαζί είναι ένα σκέτο τσίρκο. Ναι, αυτές τις ε, καταγγελίε, λέει η πρόεδρο, θα πρέπει να τι απευθύνουμε στον κατάλληλο χρόνο και στο κατάλληλο μέρος. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλουμε κάτι άλλο να ρωτήσουμε. Η ΕΚΟ μάλλον θέλει να πει κάτι για τον προπολογισμό τον ανθρωπιστικό. Ευχαριστώ Πρόεδρε για την βοήθεια την ανθρωπιστική. οι πιστώσεις είναι απολύτως και με το πολιετές ε, πλαίσιο που είχε αποφασιστεί. Εμείς θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τα μέλη της Επιτροπής για την υποστήριξή τους, ιδιαίτερα μέσα των τροπολογιών που έχουν υποβληθεί, που θα επιτρέψει στην ΕΚΟ να παρακολουθήσει και τις δεσμεύσεις του Επιτρόπου Στυλιανίδη για την παιδεία και την αφιέρωση του, μάλλον την αύξηση από 1 σε 4% των δεσμεύσεων για την παιδεία. Τώρα κατά τα άλλα ξέρετε ότι είχαμε μια πολύ ευαίσθητη κατάσταση τελευταία χρόνια, αλλά χάρη στην υποστήριξή σας, σύμφωνα και σύμφωνα με τις παρούσες ε, προτίσεις ε, που ε, μιλούν για μεγαλύτερο ποσοστό δεσμεύσεων, νομίζω ότι θα μπορέσουμε να εκπληρώσουμε απολύτως τις υποχρεώσεις μας σχετικά με αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ. Αυτό σημαίνει ότι είχαμε, έχουμε το ίδιο πρόβλημα που είχαμε και το περσινό έτος. Οι αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές δεν είναι στο ίδιο επίπεδο. Και ευχαριστούμε τους συναδέλφους που άσκησαν πίεση από πλευρά της Επιτροπής μας. Οι πληρωμές είναι πιο υψηλές από ότι οι αναλήψεις υποχρεώσεων. Μάλιστα. Δεν, το, δεν βλέπω κανέναν άλλον να πάρει να το λόγο. Α, από την Τεύκο θέλετε να πάρετε πάλι το λόγο. Ναι. Για την Τεύκο να ευχαριστήσω τον εισηγητή και τα μέλη της Επιτροπής ΔΕΒΕ σχετικά με το σχέδιο προεπολογισμού και για τις δεσμεύσει ε, και για τις πληρωμές. Για τις πληρωμές από το 2013 έχουμε μια σημαντικότατη έλλειψη, έλλειμμα και σήμερα ήδη αυτή τη στιγμή έχουμε εξοδεύσει το 80% των δεσμεύσεων ιδιαίτερα για θέματα ασφάλειας τροφίμων και περιβάλλοντος. Εκτιμούμε ότι φέτος θα έχουμε μη πληρωμένα τιμολόγια για ύψους 623 εκατομμυρίων ευρώ. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε κάθε προσπάθεια για να αποφύγουμε νέα τέτοια κατάσταση και θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και πάλι την Επιτροπή για την ε, υποστήριξή της. Σας ευχαριστούμε πολύ. Συνάδελφοι, μάλιστα, δεν ε, ζήτησε κανείς άλλος ε, το λόγο, άρα θα κλείσω και το 6. Να περάσω στα 7, στα διάφορα. Θέλει κανείς τίποτα να πει στα διάφορα. Έχει κανείς καμιά ανακοίνωση, αν όχι. Επόμενη συνεδρίαση στις 21 Σεπτεμβρίου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστή η πρόεδρο Ευγενικά και τη Εμείς σας ευχαριστούμε και καλό σας απόγευμα.